η τοποθέτηση. Πρώτο θέμα της κυρίας Μεζάρος. Δύο λεπτά. Έχει το λόγο ο εισηγητής κύριος Μεζάρος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για, την, ε, για το καλή Δεν είμαι σύντομος. Η, η, η έκθεση για την άδεια προσχώρηση ε, στο πρωτόκολλο τη ε, Σύμβαση Βιέννη δεν συζητήθηκε στην Ολομέλη και αυτό θέλω να σα ενημερώσω για το θέμα και το σκοπό τη έκθεση. Η πρόταση μα επιτρέπει να γίνουμε συμβαλόμενα μέρη τη Σύμβαση τη Βιέννη για την αστική ευθύνη πυρηνικών ζημιών και εγκρίνοντα ή προσχωρώντα στο, πρωτόκολλο. Η απόφαση του Συμβουλίου απευθύνεται στα κράτη-μέλη τη Ένωση που είναι συμβαλόμενα μέλη στην Σύμβαση της Βιέννης, αλλά δεν έχουν κυρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει το, την ε, επικύρωση του πρωτοκόλλου του 77. Οι χώρες αυτές είναι Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία. Η τροποποίηση της Σύμβασης της Βιέννης είναι η ενημέρωση των κανόνων για την ενίσχυση του δικαιώματος δίκαιης αποζημίωσης σε περίπτωση πυρηνικών ατυχημάτων. Η προσχώρηση στην, στο πρωτόκολλο του 1997 είναι θετική γιατί βελτιώνει την αποζημίωση των θυμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση του Συμβουλίου προτείνει να επιτραπεί η, επικύρωση ή η σύναψη του πρωτοκόλλου του 1997 για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Με βάση τη, σύμβαση, τη συνθήκη της Ένωσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο. Ως εισηγητής συστήνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη για να επιτρέψει τα συμβαλόμενα μέρη να συνάψουν το πρωτόκολλο του 97. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε το σχέδιο. Ποιοι είναι υπέρ. Και κόντρο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Έκθεση ποιητικά είναι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Μαρινέσκου. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ζαντό. Υπέρ. Δεν υπήρχε ονομαστική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Στον εισηγητή, συγγνώμη. Μου λένε από, ότι υπήρξε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την ε, προηγούμενη ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη. Επανερχόμαστε και ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την έκθεση Ζαντό. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. ζήτησε το λόγο πριν την ε, ψηφοφορία για την έκθεση Βίξνου ο κύριος Γκόλνης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να κάνω μια παρατήρηση πριν ψηφιστεί η έκθεση Βίξτρομ για την άρση της ασυλίας ε, της Μαρίν Λεπέν ότι η ενδιαφερομένη δεν μπόρεσε να λάβει το, να, να, να επιτύχει το αίτημά της να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια και δεν, μπορεί να, δεν μπόρεσε να παράσχει εξηγήσει για το θέμα αυτό στο σύνολο των συναδέλφων και δεν μπόρεσε για το θέμα αυτό να λάβει ώστε όλοι να έχουν την ευθύνη τους ονομαστική ψηφοφορία. Με άλλα λόγια η διαδικασία αυτή μοιάζει περισσότερο με μια διαδικασία του ανώτατου Σοβιέτ της ε, παλιάς Σοβιετικής Ένωσης παρά ενός Δημοκρατικού Κοινοβουλίου. Κύριε Γκόλνης, η διαδικασία προβλέπει η συζήτηση να γίνει στα πλαίσια της νομικής επιτροπής. Ούτω και γένετο. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα λοιπόν εναντί της συναδέλφου κυρίας Λεπέν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγνερ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σίμψον. Υπέρ. Πρώτη ομάδα τροπολογιών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η πρώτη ομάδα. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Έχει την ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια προς τον συνάδελφο κ. Σίμψον. Σάβισα Τόμαστ. 11 τροπολογίες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρόταση συνολικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Σίμψον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την έκθεση αυτή και τις εκθέσεις ε, Εντάξει, Λόβερ, θέλαμε να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Θέλαμε να αναβληθεί η ε, απόφαση για το ε, ψήφισμα, νομοθετικό ψήφισμα και να αναπευθεί το θέμα αυτό στην Επιτροπή Τουρισμού για να πετύχουμε ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε την πρόταση Σίμψον. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση Σίμψον. λόγο. 61 τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρχεται ψηφοφορία. Υφίσατε όλοι υπέρ της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επτά απολογίες Επιτροπής Μεταφορών υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. 75 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το 2, τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνολικά για την πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Σίμψον έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, και πάλι το ίδιο αίτημα με την προηγούμενη έκθεση να παραπεμφθεί στην Επιτροπή ε, Τουρισμού για να καταλήξουμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης με το Κοινοβούλιο. Ζητώ αναβολή της ψηφοφορίας του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Κούν. 102 τροπολογίες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 111. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Ωραία, ωραία. Ψηφίζουμε ο ε, έλεγχος για την 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 113. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 117. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 117. Άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσετε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 115. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επτά, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεν σηκώνετε πια το χέρι σας. Τι να κάνω. 116. Υπέρ. Κατά. Τσεκ. Για το 116 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ο κύριος Σίμψον πρόεδρος της Επιτροπής έχει το λόγο. Για τρίτη και τελευταία φορά ζητώ από το Κοινοβούλιο να αναβάλει την ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα, να ε, παραμεθεί το θέμα και πάλι στην Επιτροπή για να δοθεί η δυνατότητα διαπραγματεύσεων για συμφωνία πρώτη ανάγνωση. Ποιο ψηφίζει υπέρ τη πρόταση Σίμψον. Όχι, αποχές. Πήρε και το τρίτο του νέου κύριο Σίμψον. Έκθεση Ζίβερ. Ζέμπερ. Πρώτη ομάδα τροπολογιών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Υπέρ της προτάσεως κατά αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού, ψηφίσματος. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Έκθεση Ντόρφμαν, 21 τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 25. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίζατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ, αλλιώς υπέρ του 23 κατά αποχές. Νομίζω ότι η ίδια πλειοψηφία με πριν είναι, αλλά κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο για την 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η τροπολογία 5. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση συνολικά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Δανέλης. Παράγραφος 17. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη συνολικά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τόια. Πρώτο τμήμα παραγράφου 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Πρώτο τμήμα. Ζητήσετε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Τις 6. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται για δύο ψήφους. Ωραία. 15. 12 διορθώνει ο μιλητή. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. 15. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα γίνει έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 26 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 30 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 34 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Πρόταση συνολικά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Τόια. Μπαρτολότσι. Τροπολογία 7. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 33, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 40, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 43, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συνολικά η πρόταση, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Buon appetito. Καλή σας όρεξη. E Φύγετε σιγά σιγά αγαπητοί συνάδελφοι, ηρέμος και ησύχος, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στις ε, επεξηγήσεις.